Καλησπέρα σας. Ε, Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν σχόλια σχετικά με τα πρακτικά αυτά. Όχι, συνεπώς εγκρίνονται τα πρακτικά. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι σήμερα το απόγευμα είναι η ώρα των ερωτήσεων με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολουθούμε τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή οι ερωτήσεις διαρκούν ένα λεπτό, απαντήσεις ένα λεπτό και αν υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση 30 δευτερόλεπτα και απάντηση 30 δευτερόλεπτα. Πρώτα απ' όλα, οι επικεφαλείς, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων ε, θα λάβουν το λόγο. Πρώτον έχουμε το Coin von εξ ονόματος ε, της, ε, του ΕΛΚ. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα, πρόεδρε Μπαρόσο, να σας θέσω μία ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη την οποία επισημάνατε στη συζήτηση αυτή για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει η επέκταση του Ταμείου, η διεύρυνση του Ταμείου και πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το Ταμείο και σε ποιο χρονικό, ε, σε ποια χρονική διάρκεια Ποιο είναι λοιπόν το όραμά σας για τη διεύρυνση αυτού του Ταμείου. Thank you Ευχαριστώ. Το πολύ κύριε Μπαρόζο. Ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Ήρθατε και σήμερα το πρωί. Στην κυρία Κόριν Βόκενκούλ, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο η θέση μου και η θέση της Επιτροπής. Είναι σε αυτό το έγγραφο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δυνατότητες ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ε, πρέπει να διευρυνθεί. Είναι μέρος μιας περιεκτικής, μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και αντίδρασης. Υπάρχει μόνο μία φράση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για εξυγίανση, είναι σημαντικό για την σταθερότητα της Ευρωζώνης να αυξήσουμε τις δυνατότητες, διότι όπως ξέρετε ε, το Ταμείο έχει 440 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το ανώτατο όριο τώρα, αλλά ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν μπορεί να δανείσει τα 440 αν χρειαστεί Λοιπόν, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι βεβαίως να αυξήσουμε την χρηματοδοτική ικανότητα του Ταμείου. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ επικοδομητική πρόταση που θα πρέπει πολύ γρήγορα να υιοθετηθεί ως μέρος μιας αντιμετώπισης ολοκληρωμένης περιεκτικής. Ευχαριστώ. Υπάρχει πρόσθετη ερώτηση. Μία ερώτηση λέτε ότι καλύτερα να γίνει αυτό πιο γρήγορα και να μην καθυστερήσει. Τι εννοείται ακριβώς. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Γιατί υπάρχει φυσικά ένας χαρακτήρας καταπήγοντος. Ένας κατεπήγον ε, χαρακτήρας σε ό,τι αφορά και την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οποία θα πρέπει να επανέλθει και σήμερα βλέπουμε ότι κυρίως γίνονται συζητήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων και των υπουργών ε, οικονομικών. Πότε λοιπόν είναι αυτό το σύντομα. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος. Ευχαριστώ. Σύντομα, όχι αργά, αυτό σημαίνει ότι είδαμε στο παρελθόν ότι πάρα πολλές αγορές θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη δεν αντιδρά αμέσως. Δεν... Γι' αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες. Ε, χθες υπήρξε, συναντήθηκε η, το, η Ευρωομάδα και η το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και νομίζω ότι θα ήταν ε, ε, φρόνιμο εφόσον έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό από τις αρχές Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στίβεν Χιούς εκ μέρους ε, ε, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, πρόεδρε Μπαρόσο, ξέρω ότι υπάρχει αντίδραση για την ανάμειξη της Επιτροπής στην αγορά εργασίας της Ιρλανδίας, αντίδραση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Πάρα πολλοί ζητούν αναθεώρηση των ρητρών τιμαριθμοποίησης, αναθεώρηση των επιδομάτων και της υπερβολικής προστασίας των εργαζομένων. Η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να προωθήσει έναν διάλογο κοινωνικό και να μην υπονομεύει το θέμα αυτό και εφόσον αυτό αποκλείεται από το κοινωνικό κεφάλαιο της συνθήκης, τι νομική βάση χρησιμοποιεί ε, η Κομισιόν για να παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις αυτές τις συλλογικές. Επίσης ε, δεν ξέρω τι γίνεται με την δυνατότητα για να επιτευχθεί η διαδικασία 2020. Ποια είναι η απάντησή σας. Χωρίς αμφισημία μπορώ να πω ότι υποστηρίζουμε τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει όμως να γίνει αυτό και σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι ευθύνη των κρατών, των κρατών μελών. Προωθούμε ενεργά τον κοινωνικό διάλογο με επιχειρήσεις και με άλλους εταίρους. Αλλά Είμαστε της γνώμης ότι θα πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε περισσότερα κίνητρα για εργασία. Πρέπει βεβαίως να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας ε, και πρέπει ε, να αυξηθεί αυτό που είναι σημαντικό, η ανταγωνιστικότητα. Πρόσθετη ερώτηση. Ευχαριστώ. Γιατί, Πρόεδρε, εστιάζουμε την προσοχή μας στην αγορά εργασίας τι θα κάνουμε με την χρηματοπιστωτική αγορά, την αγορά αγαθών, την εσωτερική αγορά. Γιατί η πίεση γίνεται ως προς την αγορά εργασίας. Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι να επομίζονται το κόστος αυτής της κρίσης ή ύφεσης. Ε, όχι, λυπάμαι, απάντηση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Αναφερόμαστε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Γίνεται συντάσσετε μια ετήσια έκθεση για να το δούμε εις βάθος το θέμα. Τώρα ασχολούμαστε με την αγορά ενέργειας, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την αγορά εργασίας για να αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα για τις χώρες που είναι πιο ευάλωτες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερχόφστατ, εξ των Φιλελευθέρων. Γνωρίζω ότι μιλώντας κατηδίαν με τον πρόεδρο Μετβέντεφ μιλήσατε για τις ανησυχίες σας για την υπόθεση Κοντορνόφσκι. Δηλαδή, αν πρόκειται για μία δοκιμή για το κράτος δικαίου στη Ρωσία, τότε απέτυχε. Στις 31 Δεκεμβρίου ο Μπόρις Νέμσοφ φυλακίστηκε, συνελήφθη και δυνάμει του άρθρου 31 του συντάγματος θα πρέπει να, ε, υπάρχει, να, αντιταχθεί κάποιος αυτή τη διαδικασία και κάθε 31 του μηνός, 30 του μηνός κάθε μήνα ε, διοργανωνόταν μία διαμαρτυρία. Τώρα η διαδικασία συνεχίζεται και το 2011. Αυτό σημαίνει ότι το 2011 μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία όπως άρχισε με τον κύριο Νέμσοφ. Ποια είναι η κοινή δράση που μπορείτε να προωθήσετε επί του θέματος. Η Ρωσία είναι ε, μέλος του ΟΣΑ, ε, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. Θα πρέπει να μας πείτε πώς το αντιμετωπίζετε. Απάντηση. Όπως είπατε κύριε Φερχόφστατ, το θίξαμε αυτό το θέμα με τους Ρώσους εταίρους μας και αντιδράσαμε κατά των περιπτώσεων ε, Λέμπετεφ και Κοντορκόφσκι. Νομίζουμε ότι θα πρέπει ο δικαστικός τομέας να είναι αυτόνομος όπως ορίζουν και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να προωθηθεί η εταιρική σχέση μεταξύ ε, των δύο χωρών. Επίσης, το κράτος δικαίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο αυτής της πολιτικής θα προωθήσουμε το θέμα σε διάφορες συζητήσεις και στη διάσκεψη κορυφής της Βρυξέλλες θεωρούμε ότι η, η Ρωσία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δυνάμει των... της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα απλώς να σχολιάσω ότι το θέμα θα πρέπει να επιληθεί το ταχύτερο δυνατό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Αυτό αφορά τη Ρωσική Συνομοσπονδία, διότι έχουμε εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να, να παραμείνουν ως έχουν. Ευχαριστούμε, Πρόεδρο. Η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Ρωσία ο τύπος και η ελευθερία έκφρασης αποτελούν τεράστια προβλήματα αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ουγγαρία. Ερωτώ λοιπόν γιατί είναι τόσο χαλαρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό ε, της Ουγγαρίας για την ελευθερία του τύπου ε, παραβιάζει και καταπατά βασικές αρχές της Ευρώπης. Ζητήσαμε νομική γνωμοδότηση για τα κριτήρια της Κοπεχάγης σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά ε, οδηγίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UNESCO, τα η χάρτα των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και πάρα πολλά ακόμα νομικά έγγραφα. Ερωτώ λοιπόν πότε θα αναλάβετε τη δέουσα δράση για την Ουγγαρία, γιατί δεν υπάρχει ακόμα διαδικασία επί παραβάση και υπάρχουν και σχετικές, ε, ε, σχετική νομολογία στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εφαρμόσουμε και με την Ουγγαρία και με τις άλλες χώρες μέλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να γίνεται από, πολύ προσεκτικά από νομικής άποψης. Θα πρέπει να ακολουθείτε σαφής μεθοδολογία. Αυτό και πράττουμε. Χτες ενημέρωσα την Επιτροπή Λίμπε και Πολιτισμού και Έχουμε κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ουγγαρίας και σκοπεύουμε να αποστείλουμε επιστολή μέσα στην εβδομάδα προς την κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Μία πρώτη επιστολή στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν οι Ουγγρικές αρχές. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει να ακολουθηθούν σαφείς ε, αντικειμενικές ε, νομικές διαδικασίες γιατί η Ουγγαρία όπως κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας διαβεβαιώ ότι πολύ ενδελεχώς θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό. Η περώτηση της κυρίας Χάραμς θα μας πείτε λοιπόν γιατί όλα τα τεκμήρια που έδωσε η Ουγγρική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν διατίθενται και στο Κοινοβούλιο για να τα κοιτάξουμε και εμείς, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχει υποβληθεί το πλήρες κείμενο του νόμου και έτσι χρονοτριβούμε. Χορηγήστε μας λοιπόν, διαβιβάστε μας τα έγγραφα αυτά και να πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασκείται πολιτική, για παράδειγμα στις ε, διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και να τονίζουμε και να υπογραμμίζουμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης και να τα ξεχνάμε τα κριτήρια αυτά όταν μια χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Απάντηση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Φυσικά απαντούμε ε, στο Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, κυρία Νελικρούση ήταν χτες... Ε, η Αντιπρόεδρο Κρού ήταν χθε στι επιτροπέ του Κοινοβουλίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ακολουθείτε με αντικειμενικό τρόπο ο, η μέθοδος. Έχει πολύ καλή αξιοπιστία και πολύ καλή φήμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τέτοια ζητήματα και δεν θέλουμε φυσικά να την διακυβεύσουμε. Σα διαβεβαιώ ότι ακολουθούμε αυτά τα ζητήματα αυτά και έχουμε εκφράσει ανησυχίες. Έχω προσωπικά κατηδίαν εκφράσει ε, τις αμφισβητήσεις μου, τις αμφιβολίες μου με το, στον, ε, στον ε, κύριο Ορμπάν. Αύριο θα παρευρεθεί εδώ πέρα και θα μπορέσετε να τα συζητήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο, ο κύριος ε, Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές ημέρες η Επιτροπή ε, μια επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα αίτια της καταστροφής του Σμόλενσκ ε, στις 10 ε, Απριλίου. Το κοινό στην ε, Πολωνία εξεπλάγει από τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της έκθεσης ε, και σκέφτηκε ότι η έκθεση αυτή είναι μεροληπτική. Τις τελευταίες μέρες αποδείχθηκε ότι η έκθεση ε, καλύπτει και αποκρύπτει ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι δυσμενή για την Ρωσία και μετατοπίζει την ενοχή στην, προς την πολωνική πλευρά. Έχουν γίνει σφάλματα ε, ίσως από την δική μας πλευρά στην προετοιμασία ε, της επίσκεψης ε, του Πολωνού Προέδρου. Παρόλα αυτά η έκθεση αποτελεί αν θέλετε μια συνωμοσία και αποκρύπτει ε, στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν ε, την ρωσική πλευρά. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η ε, Επιτροπή, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα του όπου πέθανε αρχηγός κράτους όπως και μέλη της πολωνικής ελίτ. Ευχαριστώ. Κύριε Καμίνσκι, Κανείς δεν θα ξεχάσει αυτήν την τρομερή τραγωδία στην Πολωνία ή αλλού. Λυπηθήκαμε πολύ για τον θάνατο του Προέδρου Κασίνσκι και για όσους βρήκαν τραγικό θάνατο. Βεβαίως γνωρίζω την έκθεση και τις αντιδράσεις της πολωνικής πλευράς και κατανοώ πλήρως την αντίδραση λόγω της σημασίας αυτής της τραγωδίας αλλά η Κομισιόν μπορεί να δράσει μόνο όταν έχουμε τη νομική βάση να δράσουμε. Ε, ποτέ οι πολωνικές αρχές δεν μας ζήτησαν να παρέμβουμε σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά βεβαίως είμαστε πάντοτε έτοιμοι και διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε περίπτωση που θα υπάρξει ένα τέτοιο αίτημα. Αν κατάλαβα σωστά κύριε Πρόεδρε, επειδή μέχρι τώρα η πολωνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υποβάλει αίτημα τότε θα δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατάλαβα καλά. Όπως είπα θα πρέπει ε, να δούμε ε, την απονομικής πλευρά στο θέμα. Νομίζω ότι ήταν μια ε, στρατιωτική πτήση, μια επίσημη επίσκεψη και ο κανονισμός στέθηκε σε ισχύ μόνο μετά από την τρομερή αυτή τραγωδία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, έχει πολλά επιχειρήματα, έχει βάση ε, για να παρέμβει η Κομισιό, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε με τις πολωνικές αρχές αν μας το ζητήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Λόταρ Μπίσκι από την ΚΟΕ. Κύριε Μπαρόζο, όλοι γνωρίζουμε τη συμφωνία, την σημασία της σταθερότητας του ευρώ. Έχω λοιπόν κάτι που δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη συζήτηση για την ε, διεύρυνση του Ταμείου Διάσωσης ε, και εσείς, ε, εσείς μάλλον είπατε να προχωρήσουμε και η κυρία Μέρκελ είπε stop. Ερωτώ λοιπόν, δεν έχετε καμία επικοινωνία και συνεννόηση. Μπορεί αυτό να συμβεί κάποια φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο και ξέρετε αυτό τραβάει την ε, προσοχή των ε, μέσων. Είναι πραγματικά πολιτικό θέμα, δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί να σας βρει αντίθετους με την ε, κυρία Μέρκελ. Καταλαβαίνω, γιατί και εγώ δεν σύμφωνο πάντα με την κυρία Μέρκελ, αλλά εδώ το θέμα είναι μήπως ε, τελικά βοηθάμε τους κερδοσκόπους με, τη δημιουργία τέτοιας ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση κάθε κυβέρνηση έχει τις ευθύνες της ε, και καθένας πρέπει να παρουσιάζει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα πολύ συνεκτικό και πρακτικό έγγραφο εκφράσαμε την θέση μας. Αυτό δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και χρέος μας. Αυτό λοιπόν κάναμε και αυτό νομίζω ότι το δέχτηκαν πολύ θετικά οι αγορές. Το είδαμε αυτό, γιατί τώρα κατάλαβαν ότι υπάρχει πλέον θέληση να προχωρήσουν τα πράγματα, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι ομόφωνη η ανάλυση των αγορών ότι χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Αυτό ξέρετε δεν είναι μόνο θέση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της, ε, των ε, συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπαρόσο, συμπληρωματική ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι εκφράζετε τη γνώμη σας και την τοποθέτησή σας, αλλά πώς είναι δυνατόν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα το σαν θέμα που υπάρχει καρδοσκοπία εις βάρος του ευρώ σε μια τόσο χρονική, ευαίσθητη χρονική συγκυρία, πώς είναι δυνατόν να φαίνεται ότι υπάρχει διχόνοια μεταξύ ε, ημών και της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σαρκοζή. Πώς είναι δυνατόν να φαίνεται ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Απάντηση. Δεν χρειάζεται να τα κράτη-μέλη να ζητούν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού εκφράσουν τη γνώμη τους. Η πρότασή μας έγινε, ε, αν θέλετε, ακολουθώντα και τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου, όπου τα κράτη-μέλη αποφάνθηκαν ότι θέλουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εγγυηθούν την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα και αναφέρθηκαν ειδικά και στο Ταμείο και είπαν ότι θέλουν να το ενισχύσουν. Δεν υπάρχει και οποιαδήποτε αντίφαση, δεν μπορώ να σχολιάσω λοιπόν αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να πω ότι αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ομόφωνη θέση και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι ειδικά ζητήματα για το πώς επικοινωνούμε. Ευχαριστώ κυρία Μαρθά σαν λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μπαρόζο, την προηγούμενη εβδομάδα ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου που υπηρέτησε το ελεγκτικό για 15 χρόνια αναφέρθηκε στην έλλειψη ανεξαρτησίας του λογιστικού αυτού σώματος ως προς την τη δήλωση αξιοπιστίας. Η επιστολή Γκούρντα στην ουσία επιβεβαιώνει τις εξουσίες και αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής έναντι αυτού του οργάνου, τη στιγμή που χορηγείται απαλλαγή εδώ και 15 χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας εξωτερικός έλεγχος εκτός θεσμικού πλαισίου δεν μπορούμε, δεν μπορεί κανείς να απαλλάσει την Ευρωπαϊκή Επίτροπη συνέχεια. Εσείς κύριε Μπαρόσο θα επιτρέψετε έναν εξωτερικό έλεγχο αναθεώρησης των λογαριασμών για να δούμε πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Μπαρόσο. Όπως ξέρετε το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένα εξάρτητο όργανο. Εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή ως προς τους ελέγχους ή τις προτεραιότητες. Ούτε θα θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ε, είναι προς δικό μας συμφέρον να υπάρχει ανεξαρτησία αυτού του σώματος. Ποτέ δεν είχα προβεί σε αρνητικό, ε, αρνητικό σχόλια σε αρνητικό σχόλιο σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο, το 10 ή οποιαδήποτε άλλο όργανο. Πρόκειται για μία βασική αρχή της δημοκρατίας. Άρα υπάρχει διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την χάνει του ελέγχου. Και αυτό, αυτός ο διάλογος έχει μία σταθερή βάση με βάση τις ε, διεθνείς προδιαγραφές και έχουμε δεχτεί πολλές επικρίσεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό θα πρέπει να δεχτούμε την ανεξαρτησία των οργάνων και ιδιαίτερα του ελεγκτικού. Ευχαριστώ κύριε Παρόσο, διαφωνώ με την απάντησή σας. Απαντώντας στις επικρίσεις ε, του ελεγκτικού τα τελευταία δέκα χρόνια, η Επιτροπή στράφηκε στους ελεγκτές ζητώντας να αλλάξουν τη μεθοδολογία εργασίας έτσι ώστε η έκθεση για τις κοινοτικές δαπάνες να παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα. Στα πλαίσια της 30 ετούς πείρας μου ποτέ δεν άκουσα ο ελεγχόμενος να επιβάλλει στον ελεγκτή πώς θα τον ελέγξει. Πώς ξέρουμε ε, για το κατά πόσο η θέση του ευρώ σχετίζεται με μια διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί το ελεγκτικό. Απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, μπορεί να εκφράσει μια οποιαδήποτε γνώμη για τη διαδικασία ελέγχου. Αυτό κάνετε και εσείς τώρα. Εμείς ε, έχουμε εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό θα πρέπει να εκφράζουμε, να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας. Αυτό δεν αποτελεί πίεση. Πρόκειται για μια άσκηση διαφάνειας. Άρα δεχόμαστε το ελεγκτικό, δεν ασκούμε καμία πίεση στο ελεγκτικό και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εφαρμόσουμε τις συστάσεις της ανεξάρτησης αυτής ελεγκτικής αρχής. Ντάνιελ Βαντερστόπ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ιερουσαλήμ είναι μοναδική αιώνια και αδιέρετη πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ θα είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση πάντα Ισραηλινό έδαφος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι περήφανη για το Ισραήλ γιατί πρόκειται για τη μοναδική ε, δημοκρατία στο Μέσο Στο αγώνα της κατά της Ισλαμικής Τζιχάτ ε, το Ισραήλ δεν προσπίζει μόνο τα δικά του δικαιώματα αλλά και όλες τις χριστιανιστικές και εβραϊκές αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υποστήριξη προς την, το Ισραήλ θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Θα πρέπει θα να αποστείλει σαφές μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την διεθνή κοινότητα. Γιατί θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, Πρόεδρο Μπαρόσο. Συμφωνείτε μαζί σας ότι η διπλωματική αντιπροσώπηση του Ισραήλ θα πρέπει να ε, μετεγκατασταθεί στην Ισραηλινή πρωτεύουσα της Ιερουσαλήμ. Είμαστε κατά ε, των ε, πρεσβειών, αλλά αν υπάρξουν πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ μόνο. Uh, Καταρχάς, ξέρετε ότι ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το Ισραήλ. Υποστηρίζουμε την ύπαρξη του Ισραήλ και όπως είπατε πρόκειται για ένα δημοκρατικό κράτος σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε πλήρως τα δικαιώματα του Ισραήλ. Εκ παραλλήλου θα θέλαμε να γίνονται σεβαστά από το Ισραήλ τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των λασμών και θεωρού, προσδιορισμού των λαών και θεωρούμε ότι η λύση είναι η λύση των δύο κρατών τα οποία θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο ε, υπό το κράτος δικαίου. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή της πρωτεύουσα, ε, η εκπροσώπηση, η αντιπροσωπία μας ε, στο Ισραήλ δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει, να, να μεταεγκατασταθεί. Ευχαριστώ ε, συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, Πρόεδρε, με απογοητεύει η απάντηση. Ξέρετε, σας ερω... διαρωτούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ε, άδειες οικοδόμησης ε, Ιερουσαλήμ. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνουν διακρίσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ γιατί η πόλη είναι ενιαία, υπάρχει ένας δήμος. Τι λέμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι Ισραηλινές αρχές με τους ε, Ισραηλινούς που ζητούν άδειες οικοδόμησης στη χώρα τους, στην πόλη τους. Απάντηση. Θεωρώ ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εναρμονισμένη με αυτή της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά τους επικισμούς. Θεωρούμε ότι ο τρόπος που ε, αντιμετωπίστηκε το θέμα των επικισμών δεν ήταν πάντα ε, ωφέλιμος για την πρόοδο της ειρνευτικής διαδικασίας. Και αυτό είναι από τους λόγους, είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε την προσωπία μας την Ιερουσαλήμ, γιατί είναι σημαντική, εξαιρετικά σημαντική η πόλη για το Ισραήλ και για όλους μας. Ας ε, δεσμευτούμε λοιπόν προς την ειρηνευτική διαδικασία, ας σεβαστούμε τα δικαιώματα των Ισραηλινών, αλλά και μην ξεχνάμε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ. Και τώρα θα περάσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Καινοτομία και ενέργεια. Δεύτερο τμήμα των ερωτήσεων του γύρου των ερωτήσεων. Καινοτομία και ενέργεια. Ο κύριος Αλέχο Βιδάλ Κουάδρας. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την καινοτομία σε διάφορους τομείς του ενεργειακού μας συστήματος ε, μπορώ να μιλήσω για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, σύνδεξης, χάση τέταρτης γενεάς, εφή δίκτυα, ανανεώσιμες πηγαίνες ενέργειας, ε, χρήση υδρογόνου σε πυλώνες ή στήλες καυσίμων, ηλεκτρικά οχήματα και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί. Οι πόροι είναι ελάχιστοι, Πρόεδρε, και πολλοί πολίτες αναρωτιούνται και ανησυχούν. Δηλαδή, αναρωτιούνται στην παρούσα δύσκολη φάση πώς θα καταφέρει η Επιτροπή να ορίσει αυτές τις προτεραιότητες. Ποιες προτεραιότητες είναι πραγματικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Δύσκολη ερώτηση και με τις προτεραιότητες. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά. Να προσθέσουμε επίσης τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση που είναι προτεραιότητα, αλλά επίσης να επενδύσουμε σε τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα, διότι υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτήν και θα πρέπει στον τομέα των ενεργειακών να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Αυτές είναι οι τέσσερις προτεραιότητες που θα ήθελα. Ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, υλοποίηση όλων των κανόνων εσωτερικής αγοράς, ενεργειακή απόδοση, τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα και να δεχθούμε κοινή προσπάθεια στην εξωτερική διάσταση. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Ευχαριστώ η κυρία ε, Γιωρομάνα Γιόρνταν Κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020. Σε πολιτικό επίπεδο συζητούμε έναν στόχο πιο φιλόδοξο ακόμα. Είναι γνωστό ότι θα πρέπει η ο ενεργειακός τομέας και άλλοι να επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο. Ποια είναι η γνώμη σας για το πώς θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να έχουμε πιο φιλόδοξο στόχο. Τι απτά μέτρα πρέπει να λάβουμε στον ενεργειακό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέτρα, τα μέτρα τα οποία τονίσατε όταν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου είναι επίσης μια παγκόσμια διαδικασία, όχι μόνο ευρωπαϊκή. Στο Κανκούν επίσης υπήρξε ένα βήμα σημαντικό στις διαπραγματεύσεις ε, κρατήθηκε ζωντανή όλη η διαδικασία αλλά δεν ήταν αρκετή από τη δική μας άποψη για να προχωρήσουμε, για να δεσμευθούμε. Ε, για στόχους θα πρέπει να ζητήσουμε από άλλους ε, τους μεγαλύτερους ε, ρηπαντές τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες να κάνουν μια παρόμοια προσπάθεια και μέχρι στιγμή δεν έχουν δεσμευτεί οι χώρες αυτές γι' αυτό πρέπει να βρούμε τον τρόπο ούτω ώστε να προχωρήσουν και οι χώρες αυτές. Ταυτόχρονα οι χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να δεσμευθούν περισσότερο θα πρέπει να δεσμευθούν και στην αρχές Φεβρουαρίου αυτό που θα προτείνω στο Συμβούλιο είναι να επιτύχουμε περισσότερα από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης, διότι βρισκόμαστε κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε ε, να βρεθούμε ε, πρέπει ε, να έχουμε λοιπόν περισσότερα ως προς την ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Μπαρόσο. Βεβαίως η ενεργειακή ασφάλεια με χαμηλό κόστος για τους καταναλωτές στο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει όλες ε, τις χρήσεις χαμηλού άνθρακα. Γι' αυτό περιλαμβάνει τον άνθρακα, τον καθαρό άνθρακα, ενώ η χρήση μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ότι θα υποστηρίξετε ε, τις έρευνες για την δέσμευση άνθρακα και αποθήκευση στο μέλλον. Βεβαίω, μπορώ να σας δώσω την διαβεβαίωση ότι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά στο τέλος τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για την χρηματοδότηση ε, για την έρευνα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε όταν παρουσιάσουμε τις πολλαπλές προοπτικές. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ενώσιμες πηγές χαμηλής χρήσης άνθρακα και να δούμε ε, τις προτεραιότητες σχετικά με την στρατηγική για το τεχνολογικό πρόγραμμα. Αυτά τα προτείνουμε για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, κυρία Φιώνα γόμ. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, φτάσει στο κάτω από το 20% σε σχέση με τον στόχο του 20% ε, ενέργειας, διασφάλιση ενέργειας και αποταμίευση μέχρι το 2020. Γιατί δεν γίνεται αυτός ο στόχος δεσμευτικός στα κράτη-μέλη. Μπαρόζο. Προσπαθούμε να το, να το προωθήσουμε το θέμα για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αποδοτικότητα της ενέργειας βρίσκεται πολύ πίσω και προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής πολιτικής έχει ενταχθεί στους στόχους για το 2020 και τα κράτη-μέλη έχουν ορίσει και εθνικούς στόχους προς υποστήριξη αυτής της πολιτικής. Με βάση τα μέτρα η αποταμίευση, η εξοικονόμηση θα είναι της τάξης του 10% μέχρι το 2020 αλλά πιστεύουμε ότι τα τελικά σχέδια θα είναι πιο φιλόδοξα. Βεβαίως θα είμαστε κάτω από το 20%. Γι' αυτό θα ακολουθήσουμε μία πολιτική δύο ταχύτητων. Καταρχήν θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ την πολιτική αυτή και θα αναθεωρήσουμε με έκθεση προόδου το καθεστώς αυτό το 2013. Αν δούμε ότι ο στόχος του 20% δεν μπορεί να επιτευχθεί, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει δεσμευτικούς στόχους για το 2020. Ο κύριος Ράινχαρτ. Ο κύριος Μπουτιχόφερ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με τα θέματα εναρμόνισης των, της τροφοδοσίας ηλεκτρικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο, ο Επίτροπος ακολουθεί μια στρατηγική την οποία θεωρώ, θεωρούμε και θεωρεί και ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας ότι θα διαταράξει την επιτυχία της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποια η θέση σας για την διατάραξη αυτή σε ό,τι αφορά την ενιαία τιμή τροφοδότησης ε, ηλεκτρού και τι θα κάνετε προκειμένου ο κύριος Οιτινγκέρ να μην χρονοτρεβεί. Θέλει το 2012 να αντιδράσει παρά το γεγονός ότι και εσείς ο ίδιος πριν από λίγο είπατε ότι σήμερα ήδη μπορούμε να δούμε ότι δεν επαρκούν οι μη δεσμευτικοί στόχοι. Πώς θέλετε να επιταχύνετε την όλη διαδικασία. Απάντηση. Καταρχάς να σας πω ότι ο Πίτροπος Οιτινγκέρ τα προτείνει. Απροτείνει αυτή την προσέγγιση και θεωρώ ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλουμε να υπάρχει σύνδεση και με άλλους στόχους, όπως η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Τούτου λεχθέντος, νομίζουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο να τεθούν στόχοι, το θέμα είναι να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Είναι καλύτερο, θεωρούμε, τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν, να θέσουν τους δικούς τους στόχους, τους εθνικούς τους στόχους και μετά αν δούμε ότι τα πηγαίνουν καλά, έχει καλός. Ιδάλλως θα προτείνουμε τουλάχιστον δεσμευτικούς στόχους. Αλλά ξέρετε σε κάποιες περιπτώσεις η επιτυχία είναι ε, πετυχάνεται καλύτερα με εθελούσιους στόχους. Αυτό έχει αποδειχτεί. Δεν, αποδει... δεν αποκλείουμε όμως κάθε άλλο να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι για κάθε χώρα, αλλά ας δώσουμε στα κρατη την ιδιοκτησία της πολιτικής αυτής για να δούμε πώς θα πάνε. Ευχαριστώ, κύριε Ρίμπιχ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στις 4 Φεβρουαρίου έχουμε την ε, Σύνοδο για την Ενέργεια. Δύο οδηγίες συζητιούνται σήμερα. Καταρχάς, ό,τι αφορά το πλαίσιο για το νερό και το Δεύτερο είναι ο έλεγχος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτές οι δύο νομοθεσίες να εναρμονιστούν μεταξύ τους. Μιλάμε για την παραγωγή ενέργειας και θεωρώ ότι οι διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούν να διαρκούν πάνω από ένα έτος. Πέντε έτη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε έτη είναι μια Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό και να είμαστε και δυναμικοί, είναι πρόθυμοι να μειώσει αυτό το χρονικό όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μετατραπεί το πλαίσιο της ε, οδηγίας για το νερό προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα θέματα τα εργοστάσια υδροελεκτικής ενέργειας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Απάντηση. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειωθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος που παίρνει η έγκριση και η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη συχνά μας ζητούν μια χάρη, μια καθυστέρηση προκειμένου να υπάρξει σωστή εφαρμογή και να μην υπάρξει ε, στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό αφορά αυτό μάλλον ε, μας αφορά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αγορά. Ότι είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί. Δεν ξεκινάμε από το 0 το Φεβρουάριο και αυτό προκύπτει από διάφορες ανακοινώσεις, αλλά υπάρχει και διαφορετική, διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί προς ε, τη μείωση του χρονικού αυτού περιθωρίου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και από τα κράτη-μέλη προκειμένου να γίνονται όλα αυτά λίγο πολύ παράλληλα για να μην υπάρχει στρέβλος στην ιστορική αγορά. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Πέρσι για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο αν, ήταν το Πανεπιστήμιο του Cambridge στην περιοχή που εκπροσωπώ ανέλαβε σημαντική εργασία για τα θέματα αυτά. Πάρα πολλά πανεπιστικά ιδρύματα και επιχειρήσεις ε, μειώνουν μέσα στα πλαίσια του ε, προγράμματος πλαισίου των 50 ε, δισεκατομμυρίων. Βεβαίως το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ γραφειοκρατικό το Κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα για μια σειρά συστάσεων για την απλούστευση αυτής της γραφειοκρατίας. Τι κάνει ε, η ε, Κομισιόν για να ε, υλοποιήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ από την περιφέρειά σας. Ελπίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας, την υποστήριξη της ομάδας σας να συζητήσουμε το πλαίσιο για τις υποχρεώσεις, τις πιστώσεις υποχρεώσεων για την έρευνα, την ε, καινοτομία στον ευρωπαϊκό τομέα. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ είναι πολύ προχωρημένο, αλλά υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια σε φτωχότερε περιοχές που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε κονδύλια. Η απλούστευση ε, των διαδικασιών για την ε, καινοτομία και σε αυτή την περίπτωση για την έρευνα. Και αυτό ε, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η καινοτομία είναι μια από τις ε, προτεραιότητες μας ε, και χαιρόμαστε που έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλων. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πόσο σημαντικό είναι για τους επιστήμονες να μην χάνουν τόσο πολύ χρόνο σε γραφειοκρατική εργασία για να συγκεντρώσουν την προσοχή τους αυτό που κάνουν καλύτερα, δηλαδή την έρευνα. Κυρία Βίλντα Φιγκερέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της χρηματοοικονομικής κρίσης, τα προγράμματα λιτότητας ε, διχάζουν περισσότερα, προβάλλουν αντικοινωνικές πολιτικές, κόβονται οι δημόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας και της ενέργειας. Εάν συνεχίσουμε με τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, τότε οι ίδιες αυτές πολιτικές και πιέσεις προς την Πορτογαλία και προς τις ε, ευάλωτες οικονομίες θα οδηγήσουν σε μια επιδείνωση της κατάστασης ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Άρα το θέμα που τίθεται είναι να δούμε ποια μέτρα θα ληφθούν για να αλλάξει η κατάσταση για να εγγυηθούμε υποστήριξη και καινοτομία σε χώρες όπως η Πορτογαλία και άλλες όπου δεν υπάρχουν ε, δημόσιες επενδύσεις, κρατικές επενδύσεις, έτσι ώστε οι βιομηχανίες να έχουν ε, πρόσβαση στην ενέργεια, αν λάβουμε υπόψη τις υψηλές ε, τιμές του εργενερικού τομέα. Ευχαριστώ. Και η κυρία Φιγκεϊρέδο γνωρίζει πολύ καλά τη θέση μας σε σχέση με τις ε, περικοπές αυτές. Είναι αναγκαίες ιδιαίτερα έναντι μιας χώρας όπως η Πορτογαλία που έχει ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος. Στο έγγραφο που μόλις δημοσιεύσαμε ζητήσαμε από τα κράτη να μην μειώσουν τις ε, επενδύσεις ούτε στην έρευνα, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στον τομέα της ενέργειας και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται με μεγάλη επιτυχία. Και αυξάνονται τα κονδύλια για την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν ε, μείζονε δυσκολίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υφίσταται αλληλεγγύη. Γι' αυτό ποτέ δεν θα κουραστώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τονίζω τη σημασία της οικονομικής και κοινωνικής ε, συνοχής, να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία για να καταστήσουμε την αλληλεγγύη πιο λειτουργική. Η κυρία Μέρκης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η καινοτομία θα αλλάξει την οικονομία μας και την κοινωνία μας και θα πρέπει να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας. Είναι μία από τις πιο ε, κορυφαίες ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε πιο συνεκτική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όλες τις γενικές ε, διευθύνσεις. Γιατί κυρίως σε μία γενική διεύθυνση σήμερα γίνονται τα πιο πολλά. Θα πρέπει να είναι πιο ολιστική η προσέγγιση όμως. Θεωρώ ότι τα ταμεία θα πρέπει να είναι πιο συμπληρωματικά και να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό ταμείο και το διαφορετικό ταμείο να συμμετέχει. Θα ήθελα να εξετάσουμε, να εξετάσετε μια μεγάλη ε, πηγή καινοτομία και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο για την ενέργεια. Κοιτάμε κυρίως τα μεγάλα ε, project. Η καινοτομία είναι σημαντική για μεγάλα project, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τα μικρά. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα θα πρέπει να δυναμώσουμε τους πολίτες και θα πρέπει να συμφωνήσω και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που ζητούν δεσμευτικούς στόχους. Ευχαριστώ. Απάντηση. Έχετε δίκιο που ανησυχείτε για το θέμα αυτό, για την έλλειψη συνεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θέλω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα με συνεχτικό τρόπο. Οι ευρωπαϊκές ε, εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία αποτελούν ένα στόχο για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συνενώνοντας ε, τέτοια project ε, σε ε, ένα κατά από μία ομπρέλα, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πανευρωπαϊκές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Άρα, ένα στόχος είναι να επιταχύνουμε τη διάρκεια που παίρνει μία έρευνα προτού αποδώσει συγκεκριμένα προϊόντα για την αγορά. Αυτό θα δημιουργήσει ε, μια πλατφόρμα συνεργασίας. Αυτό προσπαθούμε να πατήχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργασία με τα κράτη-μέλη με συνεκτικό τρόπο που θα ξεπερνάει τις γενικές διευθύνσεις αλλά και τις χώρες ίσως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαβράκο. Κύριε Πρόεδρε, επιστημονικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο διεθνή τύπο και πρόσφατα εντονότερα στον ελληνικό ισραηλινό και κυπριακό τύπο αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή του αιγαίου και νότια της νήσου κρήτης. επομένως υπάρχει ενεργειακός πλούτος στον εδαφικό χώρο στα εδαφικά όρια της ευρωπαϊκής ένωσης. με τα δεδομένα αυτά ερωτάστε κύριε πρόεδρε πώς προτίθεται η ευρωπαϊκή επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποβοηθεί στις έρευνες για την ανίχνευση και εκμετάλλευση των πηγών αυτών ενέργειας οι οποίες εν πάση περιπτώσει είναι ευχερέστερο να μεταφερθούν στην ευρωπαϊκή ένωση καλύτερα από κάθε άλλο σχεδιασμένο αγωγό. και με την ευκαιρία κύριε πρόεδρε του κοινοβουλίου και κύριε πρόεδρε της επιτροπής επιτρέψτε μου να σας δηλώσω ότι σας θεωρώ πολύ τυχερούς ανθρώπους διότι η μοίρα σας επεφύλαξε στον μεν πρώτο να προεδρεύει ενός διευρυμένου κοινοβουλίου από πλευράς αρμοδιότητας μετά την εφαρμογή της συνθήκης της λισαβόνας στο δε δεύτερο να χειρίζεται μια μεγάλη οικονομική κρίση της ευρώπης. συμμερίζομαι όλες τις κινήσεις του κυρίου Μπαρόζο ως προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα ήθελα να προτείνω κάτι. Υπάρχει και η μέθοδος της Αμερικής. έκδοση νέου χρήματος. Παρακαλώ, Uh, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Έχουμε μια, ένα μακρύ κατάλογο ατόμων που θέλουν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπαρόζο. Ναι, ήθελε κάτι να μου πει κάτι ευχάριστο. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, κύριε Σαλαβράκο. Σχετικά με το πρώτο μέρος της παρέμβασής σας, εμείς δεν έχουμε τα μέσα και δεν είναι προτεραιότητα μας τώρα να κάνουμε ε, διερεύνηση ε, και να, άλλων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Η προτεραιότητά μας είναι ως προς τις υποδομές, είναι η διασύνδεση, είναι η αγωγή, ε, διότι αυτό είναι μια κρίσιμη ευρωπαϊκή διάσταση και από αυτή την άποψη θα κάνουμε προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επειδή ήδη ε, κάτι έχει γίνει για τις βαλτικές χώρες και τώρα εργαζόμαστε με τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για να υπαρχουν υπάρχουν διασυνδέσεις βορρά-νότου και προχωρούν καλά τα πράγματα και ήρθα από το Αζερβαϊτζάν ε, για τον νέο άξονα ένα νέο τρόπο ε, μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη. Αυτό μπορούν να γίνουν εκεί μερικές επενδύσεις για υποδομή ενέργειας. Ο κύριος Άρτουρ Σκάρινς. Κύριε, Πρόεδρε Μπαρόσο, η Επιτροπή έχει ε, προωθήσει ε, πρωτοβουλίες πολύ χρήσιμες κατά τη γνώμη μου για την ενεργειακή απόδοση για τα δίκτυα τα πετρελαίου, τα δίκτυα αερίου για αυτές τις ε, διασύνδεσεις. Οι δαπάνες είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται και ε, μέχρι το 2020 υποχρεώσεις αυτές. Τα μισά θα πρέπει να προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Από ό,τι απομένει από τα 100 δις που χρειάζονται μέχρι το 2020 για τα δίκτυα, από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια, από κοινοτική χρηματοδότηση ή από ε, ομόλογα, αναπτυξιακά ομόλογα, ομόλογα έργων που θα εκδοθούν ή θα υπάρξει άλλη χρηματοδότηση. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Όπως είπατε πολύ σωστά, 200 δισεκατομμύρια επενδύσεων χρειάζονται για υποδομές αερίου ε, μέχρι το 2020. 100 δίσα από αυτά ε, θα δοθούν από μόνο την αγορά, ενώ τα άλλα 100 θα χρειαστούν ε, δημόσια δράση για την μόχλευση των αναγκαίων κεφαλαίων. Γι' αυτό προτείνουμε αποσύνδεση μέτρα ούτως ώστε να γίνει πιο ορθολογική ιδιωτική επένδυση και πιο ωφέλιμη. Επίσης θα, θα εξετάσουμε τις διάφορες πρακτικές για το κόστος στο υπόλοιπο, το υπόλοιπο κενό προτείνουμε ένα νέο μέσο χρηματοοικονομικό για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013 εκτός από επιδοτήσεις μπορεί να προταθούν ε, ε, μετοχικές ε, συμμετοχές, επίσης και δάνεια και σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν επίσης, έχουν αναφερθεί τα project bonds, ομόλογα δηλαδή για συγκεκριμένα έργα αναπτυξιακά. Η κυρία Σόνια Αλφάνο. Η Οδηγία 77 του 2000 μιλά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκεί όπου χρειάζονται και υπάρχουν ε, δημόσιες προμήθειες και γίνεται λόγος για αποτέφρωση των αποβλήτων. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς ε, είχαμε ορίσει ότι θα κατασκευαστούν αποτεφρωτές οι οποίοι όμως είναι επιζήμιοι για την ανθρώπινη υγεία. Ε, η Ιταλία έχει προσαχθεί στο ΔΕΚ με βάση δύο διαδικασίες επί παραβάση και δυστυχώς γίνεται ακόμα χρήση. Ίσως δεν θα θυμόσαστε την κατάσταση, γι' αυτό σας υποβάλλω και γραπτή ερώτηση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανανεώσιμες πηγές όταν πρόκειται για αποτέφρωση μη αποδομήσιμων αποβλήτων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η αποτέφρωση δεν είναι μια σωστή διαδικασία με βάση την, ε, διαδικασία, την οδηγία 77 κάθετος 2000. Mrs. Alfano, you uh, όπως είπατε σωστά, είναι πολύ λεπτομεριακή ερώτηση. Δεν ξέρω την όλη διαδικασία επί παραβάση. Ως προς την ενέργεια και την εσωτερική αγορά έχουμε 77 διαδικασίες επί παραβάση κατά των κρατών μελών και 55 ως προς την εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να μου υποβάλλετε το ερώτημα γραπτό σας παρακαλώ για να σας απαντήσω. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καινοτομία, η προστασία του κλίματος, η στρατηγική της Ευρώπης του 2020 θα θεωρούσε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαρή σε ό,τι αφορεί το περιβάλλον και τα ενεργειακά μέτρα, αλλά πέρα από τον τίτλο αυτό κρύβεται μια άλλη ενεργειακή στρατηγική ε, η πυρηνική ενέργεια η οποία λέγεται ότι είναι καλή για το περιβάλλον και αναφέρθηκε από την Επιτροπή ότι η πυρηνική ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στην, στον ενεργειακό πακίτο και θα συνεχίσει να το πράττει αυτό. Αυτό κυρίες και κύριε, 25 χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ. Ερωτώ λοιπόν Πρόεδρε, θεωρείτε κι εσείς ότι όντως με καθαρή τη συνείδηση μπορούμε να πουλήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες την πυρηνική ενέργεια ως μια καθαρή περιβαλλοντικά ενέργεια. Ευχαριστώ. Ξέρετε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Σεβόμαστε ε, πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Κάποια κάτι μέλη τη χρησιμοποιούν, κάποια άλλα όχι κανείς δεν ε, εξαναγκάζεται να χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια, αλλά είναι αληθές ότι σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος είναι λιγότερο ρηπαίνουσα η μορφή αυτή η ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια του τουλεχθέντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες ε, υποχρεώσεις υπό τη συνθήκη της ε, Euratom. Στην αρχή υπήρχε η κοινότητα Euratom και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον να παρέχει στα κράτη-μέλη ένα σύστημα το οποίο παρέχει ασφάλεια σε τέτοια θέματα. Και αυτό λοιπόν αποσκοπούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βόλσκι. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, αναφέρατε Μάλλον μα αποστέλλεται ε, από το Αζερμπατζάν και το Τουρμενιστάν ένα αισιοδόξο μήνυμα ότι το μοναδικό πρόβλημα είναι τα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν μπορέσατε να φτιάξετε τα αριθμητικά στοιχεία αυτά με το Αζερμπατζάν και το Τουρκμενιστάν σε ό,τι αφορά τους, τα εκατομμύρια τόνων ε, αερίου. Υπάρχουν όμως ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποια απάντηση για τον νότιο διάδρομο και τον αγωγό Ναμπούκοφ που υποτίθεται ότι θα μας παρέχει ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα αέριο απάντηση από την επίσκεψη αυτή στο Αζερβαϊτζάν και στο Τουρκμενιστάν ήρθα με μια σαφή δέσμευση και των δύο χωρών να υποστηρίξουν πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον νότιο διάδρομο. Υπέγραψα μια κοινή διακήρυξη με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, τον κ. Αλιεύ, και δημόσια ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν ο κ. Μουαμέντοφ δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να παρέχει, να προμηθεύσει ε, παρκές αέριο για την Ευρώπη. Ακόμη και παραπάνω ποσότητες από αυτές που χρειαζόμαστε σήμερα. Ωστόσο υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Κάποια προβλήματα είναι οι εμπορικές αποφάσεις των εμπλεκομένων εταιριών και ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι αγωγοί μπορούν να κατασκευαστούν και να αναπτυχθούν. Υπάρχει όμως επαρκές αέριο στην περιοχή προκειμένου να προμηθευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μελη μπορούν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεργαστεί με τα κράτη αυτά είτε μέσω το πρόγραμμα Ναμπούκοφ είτε με άλλους αγωγούς. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση κύριε Τσικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει κυρία Τσικάου και διακόπτη. Βλέπουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές οικογένειες επειδή αυξάνεται η ανεργία ε, καταβάλουν πάνω από το 10% των εισοδημάτων μηνιαίως για να πληρώσουν τις διάφορους λογαριασμούς, ιδιαίτερα του ηλεκτρικού. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Λαμβάνεται υπόψη και τη συμμετοχή του ΕΤΠΑ σε αυτή τη διαδικασία, να το χρησιμοποιήσουν δηλαδή τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές ανάγκες αρχίζοντας από τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Η ε, εσωτερική αγορά ενέργειας ορίζει υψηλές προδιαγραφές ε, αντιμετώπισης και δίνει επιλογές στους καταναλωτές. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους τομείς όπου προτείνουμε ε, μέτρα που στοχοθετούν τον καταναλωτή. Ως προς την ε, καταβολή του αντιτίμου για λογαριασμούς ε, ηλεκτρισμού ή ενέργειας, πιστεύουμε ότι η ενεργειακή αγορά μπορεί να επιτύχει περισσότερα από την παρούσα κατάσταση, όπου υπάρχουν αρκετές ε, δυσλειτουργίες και κατοχή δεσπόζουσας θέσης ορισμένων επιχειρήσεων θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβάλλουμε ένα σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Δηλαδή, πολλά θα προέλθουν από τις αγορές της ίδιες, αλλά και από τις κρατικές επενδύσεις, όπως θα προβάλλουμε μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συζήτηση ως προς το θέμα της καινοτομίας και ενέργειας. Και σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής που παρευρίσκεστε εδώ για δεύτερη φορά σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.